Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Καθίστε παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να κήρυξουμε την έναρξη αυτής της ε, μεικτής συνεδρίασης, κοινή συνεδρίαση Επιτροπής Προπολισμών και Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συμπροεδρεύσω από τον κύριο Φέρμπερ, αντιπρόεδρο τη Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, γιατί ο κύριος Γκουαλτιέρη δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί θέμα της συνεδρίασής μας είναι η παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Κύριε Φέρμπερ, έχετε να κάνετε σχόλια πριν δώσουμε το λόγο στους συνεισηγητές. Πολύ σύντομα, αν μου επιτρέπετε, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρήκαμε ημερομηνία, αγαπητοί συνάδελφοι, για την κοινή αυτή συνεδρίαση από ό,τι γνωρίζω ήταν κάπως δύσκολο. Είναι όμως κάτι που έπρεπε να γίνει και χαίρομαι πολύ. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε δίνοντας αμέσως το λόγο στους δύο εισηγητές. Καθένας έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά. Ο Ούντο είναι στη δική μου λίστα ο πρώτος ε, στον κατάλογο. Ε, μπορώ να προσφέρω την τη σειρά μου στον κύριο Φερνάντε. Μετά από το συνέδριο της ε, χώρας σας, ε, του κόμματος σας στη χώρα σας πρέπει να είστε σε καλή φόρμα, λέει ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δείτε <coughs> τη δυνατότητα να συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, χαίρομαι που βρήκαμε χρόνο για να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων 2 Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεισηγητή μου, τον κύριο Μανουέλ, Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες, με τον οποίο, όπως και με το πρώτο εύση, ε, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και έχουμε λοιπόν τώρα να σας παρουσιάσουμε μία ε, πρόταση την οποία θα μπορείτε να τροποποιήσετε με τις τροπολογίες σας για να ε, βελτιώσετε το κείμενο εφόσον αυτό είναι δυνατό και σίγουρα είναι δυνατόν. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες, γιατί επέτρεψαν το να γίνει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά ε, όλη αυτή η εργασία. Ήδη υπάρχουν μεταφράσεις ε, σε όλες τις γλώσσες, ε, άρα όχι μόνο στα αγγλικά όπως φοβόμασταν στην αρχή, αλλά ο καθένας μπορεί να μελετήσει την πρότασή μας στη γλώσσα της επιλογής του και να καταθέσει έτσι και τις τροπολογίες του. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός Ποιο ήταν ο στόχος μας ε, σε αυτή την πρόταση. Κυρίως, όπως πάντα, ο στόχος να μειώσουμε το πνευματικό κενό στην Ευρώπη. Θέλουμε στο μέλλον να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολίτες. Πιστεύουμε πάντοτε ότι η νομοθεσία σε ό,τι αφορά το FC1 ήταν θετική, ήταν καλή, πετύχαμε τους στόχους μας. Ε, έχουμε βέβαια κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά κάποιες πρακτικές ε, στην υλοποίηση. Και με τις προτάσεις μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα κενά, τις αδυναμίες στην υλοποίηση. Ποια σημεία είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα η προσθετικότητα, ο ορισμός της αρχής της προσθετικότητας ε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βλέπουμε η προσθετικότητα να θεωρείται πάρα πολύ τεχνική. Δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατηγορία special activity. Χρειάζεται μαθηματική υπολογισμοί ε, και θεωρούνται κάποια πράγματα ε, επικίνδυνα από πλευράς ε, ότι ενέχουν κάποιο επενδυτικό ρίσκο και πρέπει να γίνουν πολύ περίπλοκοι τεχνικοί υπολογισμοί. Στο πρώτο εύση Υπήρχαν αυτά κενά. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους τομείς πολιτικής στο FC1 που είχαν προβλεφθεί με τις, ε, με τις ανάγκες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και χρησιμότητας. Θέλουμε να είναι πιο χρήσιμη νομοθεσία στο πλαίσιο του FC2. Οπότε εμβαθύνουμε και διευρύνουμε τις προτάσεις Κομισιόν. οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, έχουμε το θεματολόγιο 2030. Θα πρέπει να δούμε με βάση αυτά ποια ε, έργα και σχέδια είναι σημαντικά και ποια θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Το scoreboard επίσης ε, θέλουμε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για να δούμε ποια σχέδια και με ποια σειρά θα ε, προβλέπονται. Μπορεί στατιστικά, παραδείγματο χάρη, να θεωρείται ρίσκο η χρηματοδότηση των γερμανικών σιδηροδρόμων. Ε, υπάρχει και το clouding out για τους μακροπρόθεσμους ιδιώτες επενδύσεις που θα προέβαιναν σε κάποιες επενδύσεις και δεν μπορούσαν πάντα λαμβάνοντα υπόψη τη θεωρούμε ότι το ΕΦΣΙ σε ό,τι αφορά ε, το πιο ρηψοκίνδυνο μέρος μιας επένδυσης ε, θα πρέπει να συμμετέχει. Να δούμε τι γίνεται στις περιφέρειες όπου θέλουμε να υπάρχει αντίκτυπος, όπου δεν υπάρχουν επαρκείς οικονομικοί πόροι. Εκεί με, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις αναπτυξιακές τράπεζες, εφόσον υπάρχουν εκεί ιδιωτικέ. Ε, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ε, τους υπόλοιπους φορείς. Τουλάχιστον στο πιο ρηψοκίνδυνο μέρος της επένδυσης θα πρέπει το ΕΦΣΥ να μπορεί να αναλαμβάνει το ρίσκο. Και γι' αυτό θέλουμε στην προκειμένη περίπτωση να παροτρύνουμε σε μια αλλαγή νοοτροπίας και φιλοσοφίας ό,τι αφορά την ε, ανάλυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επίσης τον τρόπο συντονισμού του ΕΦΣΥ, πώς ε, θα πρέπει να τη διαχείριση των διαφόρων δραστηριοτήτων. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό για εμάς και θέλουμε να επανέλθουμε ε, σε αυτό που είχαμε προτείνει παλαιότερα για το FC1. Δηλαδή να, υπάρχουν, να υπάρχει συμμετοχή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Steering Board για να μπορεί να αποφασίζει και όταν δεν γίνεται αυτό έχουμε προτείνει μια άλλη δυνατότητα θέλουμε μια ε, εύρωστη πολιτική οι πλατφόρμες πρέπει να ενισχυθούν και με τους δεμεσολαβητές να είναι πιο εύκολο τα χρήματα να ε, διατεθούν στις περιφέρειες ε, και στους ε, διαφόρους φορείς. Το ΕΦΣΙ πρέπει να έχει, αν θέλετε, καλύτερη φόρμα, να βρεθεί σε μια καλύτερη φυσική κατάσταση. Και επαναλαμβάνω σε ό,τι αφορά το σκέλος της υλοποίησης στις περιφέρειες. σε ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρος Φέρμπερ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον άλλο εισηγητή, τον κύριο Χωσημανέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, κυρίως τον ε, συνάδελφο, τον Σκιώδη Συγητή. και τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων να κάνει τα πρώτα του βήματα ε, εδώ και μισή χρόνο. Ήταν ε, μεγάλη η επιτυχία του τώρα και ξεπερνάει τα όρια των καλύτερων προσδοκιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εύση δεν μπορεί να βελτιωθεί. Βεβαίω και μπορεί να βελτιωθεί. Ω προ ε, την ε, σωρευτικότητα, την γεωγραφική κατανομή, την τομεακή κατανομή. Το εργαλείο αυτό που έχει προσφέρει μέχρι και πόρους στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση 400, 450 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν ο στόχος του δεν είναι το κέρδος. Αυτά είναι όλα θετικά στοιχεία. Αλλά έχει συμβάλει και στην απασχόληση. Έχει συμβάλει στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα χάσμα, ένα gap στις επενδύσεις σε ένα τέτοιο εργαλείο είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε λοιπόν όλες τις δυνατότητες. Η πλατφόρμα υποστήριξης του επενδυτού είναι σημαντικό να ενισχυθεί. Ακριβώς για να ε, καλύψουμε αυτό το χάσμα. Χρειάζεται να προσφέρεται βοήθεια σε όλες τις περιοχές που την χρειάζονται, εκεί που πρέπει να γίνουν έργα και επενδύσεις. Η βοήθεια λοιπόν για να δημιουργηθούν καλύτερες πλατφόρμες και ω προ την ποιότητα και ω προ τον αριθμό του. Είναι σημαντικό. Θα μπορούσαν να υπάρξουν διασυνδέσει σε σημεία επαφή όπου οι εθνικέ, οι περιφερειακέ αρχέ και οι επενδυτικέ τράπεζε αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση. Ή τουλάχιστον μέχρι και παρόμοιε, παράλληλε δομέ σε εθνικό επίπεδο. Το Ταμείο αυτό δεν έρχεται να αντικαταστήσει τα κονδύλια τη πολιτική συνοχή έρχεται να λειτουργήσει επιπρόσθετα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε σε σχέση συνεργασία μεταξύ των διαθωτικών ταμείων και ε, όσων ε, κονδυλίων προέρχονται από το ΕΨΙ. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να σχεδιαστούν καλύτερα για το σκοπό αυτό. Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται μικρότερα έργα και προγράμματα που δεν θα πρέπει να παραμένουν μόνο στο ε, παρασκήνιο. Είναι σημαντικό στοιχείο η σωρευτικότητα, η προσθετικότητα. Αλλά η προσθετικότητα αυτή δεν είναι ίδια για το ίδιο έργο σε όλε τι περιοχέ. Το ίδιο έργο δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο, την ίδια προσθετικότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ούτε καν στο ίδιο το κράτο μέλο εντό το οποίο εκτελείται. Σε όλε τι περιοχέ δηλαδή αυτού του κράτου. Άρα οι επιπτώσει ε, στην απασχόληση είναι διαφορετικέ. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Κάτι άλλο σημαντικό είναι το θέμα τη χρηματοδότηση. Είναι ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία οι θεσμοί και οι φορεί να σέβονται τι συμφωνίε. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν υπογράψει να στηριχθούν τα προγράμματα Οριζόντας 2020 και ο μηχανισμός Διευκόλυνση διευκόλυνσης διασύνδεσης της Ευρώπης μέσω του ΕΦΣΙ 1 Θα πρέπει η δέσμευση αυτή να τηρηθεί, να γίνει σεβαστή. Πάκτα Σερβάντα Σούντ. Εδώ πρέπει να προσφερθούν εγγυήσεις εγγύησης ώστε το πρόγραμμα αυτό να περάσει από τα 500 εκατομμύρια ευρώ αλλά χωρίς να ανατρέξει ε, στα ε, κονδύλια του μηχανισμού διευκόλυνσης διασύνδεσης της Ευρώπης. Θα πρέπει να αναζητήσουμε φρέσκο χρήμα από τον προπολογισμό για να ενισχύσουμε ε, το Ταμείο Εγγύσεων. Και να μπορέσουμε επιτέλου να κινητοποιήσουμε, να βρούμε αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πρέπει η διευκόλυνση και τη της Ευρώπης να πληγεί από το ΕΦΣΙ και από την παράτασή του. Προτείνουμε αυτά που προορίζονταν για τα δημοσιονομικά εργαλεία, το ΣΕΦ δηλαδή, τον, ε, την διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης. να πάνε αυτά στο κεφάλαιο των επιδοτήσεων. Αυτά, αλλά θα φανούν και στις τροπολογίες μας και ελπίζουμε ως τον Ιούνιο και εμείς και το Συμβούλιο να συντονιστούμε, γιατί θέλουμε ένα νέο εργαλείο. Ένα νέο εργαλείο για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σκιώδη ηγητέ των δύο επιτροπών, έκον με σκιώδη για το έργο τον κύριο Κάρας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι σαφής ο εισηγητής, οι εισηγητές ότι όταν ε, θέλουμε να μείνουμε στη Champions League ε, των στρατηγικών επενδύσεων δεν μπορούμε να κάνουμε απλώς εξοραϊστικές παρεμβάσεις στη δεύτερη έκδοση του ΕΤΣΕ. Πρέπει να έχουμε πολύ πιο ουσιαστικές αλλαγές και πρέπει να ορίσουμε νέα ορόσημα. Και έτσι πιστεύω ότι το σχέδιο έκθεσης είναι μια καλή βάση για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Σε πολλά σημεία βαίνει προς την ορθή κατεύθυνση. Έχει και τον προσδορισμό της προσθετικότητας και την εντικοποίηση των κατευθύνσεων για τις πλατφόρμες επενδύσεων, ορίζει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για συμβουλή σχετική με επενδύσεις και φροντίζει να εξασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια κατά την επιλογή των έργων και των επενδύσεων. Και γενικά βελτιώνει τις δομές με βάση τα όσα έχουμε συλλέξει ως εμπειρία. Το έτσι λοιπόν είναι σε καλό δρόμο. Αλλά πρέπει να γίνει και η αξιολόγηση, είναι πολύ σημαντικό. Τρεις αρχές και προτάσεις έχω να προτείνω. Καταρχάς θέλουμε ποιοτικά προγράμματα να υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ, προγράμματα τα οποία δεν έχει καλύψει η αγορά με τη χρηματοδότησή της. Το σε ποιο κράτος μέλος θα γίνεται το έργο έχει σημασία για την ε, κάλυψη του κινδύνου για το έργο και ένα ζήτημα το οποίο ανέφερε και ο κύριος Μπούλμαν. Το προφίλ κινδύνου του έργου ε, είναι διαφορετικό από αυτό του προφίλ κινδύνου του ίδιου του κράτους το οποίο θα υλοποιηθεί το έργο. Και άρα μπορούμε να ή πρέπει να βρούμε ένα μέσον για να το υπολογίζουμε αυτό. Τα κριτήρια έτσι πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα, η προσθετικότητα σε σχέση με τα υφιστάμενα έργα και την πρόσθετη κινητοποίηση ε, κεφαλαίου επενδυτικού να εξασφαλίζεται. Και για να ολοκληρώσω, ε, δια... συνοριακή συνεργασία με τρίτα κράτη πρέπει να είναι δυνατή, αλλά και σε αυτό χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη στο σχετικό κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Βέμπερ, Φέρμπερ, μια και αρχίσαμε σχετικά αργά. προσπαθώ να είμαι πιο αυστηρό στο χρόνο και τον περιλούσε δύο λεπτά για τον καθένα. Η κυρία Καρσεβάλ Ρουβιάλ, ε, εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, Σκιώδης. Σε ό,τι αφορά την έκθεση για την υλοποίηση του ΕΦΣΥ και ε, αυτό που συζητούμε σήμερα, πολλές ε, ιδέες νομίζω προέρχονται και από την αξιολόγηση που κάναμε τη λειτουργία του πρώτου ΕΦΣΥ και τι είπαμε μεταξύ άλλων και τι θέλουμε να διευκρινίσουμε περισσότερο με το δεύτερο εύση. Είναι η επικοινωνία, ε, η δημοσιοποίηση αυτού του επενδυτικού σχεδίου, γιατί λίγοι γνωρίζουν τι είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο και πολύ λιγότεροι πώς λειτουργεί. Και αυτοί που ξέρουν και έχουν καταφέρει να χρηματοδοτήσουν ένα έργο τους ε, δεν έχουν ιδέα ότι πίσω από αυτό είναι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως με τις ε, ΜΜΕ, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο έργο. Ούτε καν ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πίσω από τη χρηματοδοτική ενίσχυση στη χρηματοδότηση. Επίσης, μεγαλύτερη διαφάνεια και κυρίως προσθετικότητα. Σε ό,τι αφορά την προσθετικότητα, λοιπόν. Ε, θέλουμε επίση περισσότερε πληροφορίε για το πώ επιλέγονται τα έργα, κριτήρια, scoreboard ε, και αυτή η προσθετικότητα γιατί κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουμε γιατί χρηματοδοτήθηκε κάποιο έργο. Και αυτό οφείλεται ίσως ότι δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση. Και μας δημιουργούνται αμφιβολίε. Τρίτον, Υπάρχει το Advisory Hub. Αυτοί πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο. Πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στον εντοπισμό έργων και σχεδίων. Να βοηθούν για την επιλογή ε, των κατάλληλων έργων. Και κυρίως, νομίζω το είπε ο κύριος Φερνάντες. Έργα μικρής κλίμακας. Πολλοί δεν έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό ε, το πολύπλοκο σύστημα, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς πώς να έχουν πρόσβαση. Τέταρτον, προϋπολογισμούς. Δεν θέλω όπως σε λεπτομέρειες. Δεν μας άρεσε που στην πρώτη πρόταση, το ε, πρώτο ΕΣΥ, αφαιρέθηκαν κονδύλια από το Connecting Europe και από τον ορίζοντα 2020 και φυσικά και δεν μας αρέσει να συνεχίσει ε, να αφαιρείται ε, προϋπολογισμός από το Connecting Europe. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για το θεματολόγιο του 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε. Γιατί να αλλάξουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει αυτό το στοιχείο στην πρόταση. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ. Επιτροπή όμως προς τον κατάλογό μου. Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε θα έπρεπε να πω, είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε την παράταση της λειτουργίας του ΕΦΣΥ διπλή διάρκεια ε, και οικονομική πρικοδότηση. Πολλές φορές έχει υποθεί, αλλά θα επιμένω και θα το επαναλάβω και εγώ. Το ΕΦΣΙ μπορεί να είναι ένα καλό project, μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν είναι πανάκια. Δεν καλύπτει τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε και άλλα για να έχουμε ένα καλό επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να γίνει με διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, άρση των εμποδίων για επενδύσει, με την ολοκλήρωση τη εννέα αγορά, με την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου, καλύτερη νομοθεσία, μείωση της ε, γραφειοκρατίας. Αυτά πρέπει να τα τονίζουμε. Το ΕΦΣΙ μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να τονώσει το επενδυτικό κλίμα, αλλά δεν είναι η πανάκια. Χαιρετίζουμε τις συζητήσεις για την παράταση της λειτουργίας του ΕΦΣΙ. Σήμερα έχω να πω τρία πράγματα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι συμμερίζομαι τις αμφιβολίες του Ελληνικού συνεδρίου για το κατά πόσο είναι παράταση αυτή, πως είναι κάπως πρόημη, πρόωρη. Κοίταξα και την ατζέντα μου σήμερα το πρωί. Δεν ήταν η 5η Ιουλίου του 2018 η ημερομηνία που είχαμε πει. Όχι, ήταν 5η Ιουλίου 2018, σήμερα είμαστε 20 Μαρτίου 2017. Και είδα ανακοινώνει κομισιόν ε, παράταση. Από τις 16 ε, ε, Ιουνίου, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα. Επίσης, ό,τι αυτό τον αντίκτυπο του ΕΦΣΙ, νομίζω θα ήταν καλό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, τα πράγματα τώρα είναι αυτά που είναι. Δεύτερον, υπάρχουν αμφιβολίες και εκφράζονται και στην έκθεση Ersten Young για την προσθετικότητα. Αναφέρεται εκεί τι θα γίνει με το crowding out effect και θα καταθέσουμε τροπολογίες σχετικά. Ελπίζω να συζητηθούν. Τρίτον, και τελευταίο. Στο ό,τι τη γεωγραφική κατανομή, ανησυχίες και εδώ έχω να εκφράσω. Αν δείτε το ΑΕΠ, το πληθυσμό, θα δείτε ότι είναι πολύ λιγότερο συγκεντρωμένα τα project από ότι αν λαμβάνονται υπόψη αυτά τα κριτήρια. Και θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Φερνάντε, τον συζητητή. να δούμε την προσθετικότητα, αλλά ε, πιο πολύ σε σχέση με τις περιφέρειες. Εκεί νομίζω μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Φέρμπερ. Ο Μπέρντ Κέλμερ για δύο λεπτά έχει τώρα το λόγο από την ομάδα ACR. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα και θα τονίσω ιδιαίτερος ότι μου φαίνεται κάπως ε, υπερβολικό να λέμε τώρα και διαπαντός ότι το έτσι είναι μια τεράστια επιτυχία. Χωρίς να ισχυρίζουμε ότι πρόκειται για το αντίθετο, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και τεράστια επιτυχία, γιατί τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου είναι ε, δηλωτικά μόνο του ότι έχει φέρει μερικά κάποια αποτελέσματα, χωρίς όμως θεαματικά επιτεύγματα. Ε, το ζήτημα της προσθετικότητας, το ζήτημα του εάν υπήρχε η δυνατότητα με άλλα μέσα ή άλλες πηγές χρηματοδότησης ε, να εξασφαλίσουμε ε, λύσεις καλύτερες ε, ή αν το έτσι δεν επιτρέπει ενδεχομένως να αναδειχθούν άλλες λύσεις και μέσα χρηματοδότησης είναι ζητήματα τα οποία με προβληματίζουν. Βεβαίως και το χρήμα μπορεί να οθήσει και να προαγάγει κάθε είδους επένδυση αλλά φέρνει προσθεμένη αξία το χρήμα αυτό προσφέρει κάτι στον πολίτη, εξασφαλίζει περισσότερη ανάπτυξη. Αυτό για μένα δεν είναι σαφές ακόμη. Και γι' αυτό στην τωρινή χρονική στιγμή δεν βρίσκω σκόπιμο να παραταθεί, δεν βρίσκω αποδεδειγμένη την ανάγκη να παραταθεί το έτσι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριο Φέρμπερ. Η φιλελεύθερη Τρεμόσε Ραμόν Παρσέλς δεν είναι εδώ. Ο κύριο Τόλβαλς όμω είναι εδώ. Νίλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ Ούντο και Ζωζέ Μανουέλ για την πολύ καλή σας δουλειά. Εκτιμώ τις προτάσεις να μην υπάρξουν και άλλες περικοπές στη διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης. Ως εισηγητής να πω ότι δεν θα έπρεπε να εξαλείψουμε όλες τις αναφορές στο ΣΕΦ, στο, ΕΦΣΥ, στο σχέδιο έκθεσης για το ΕΦΣΥ. Είναι ένα πρόβλημα για μένα, ίσως όχι για την Επιτροπή σας, και είναι καθήκον μου να το επενθυμίσω για να το λάβετε υπόψη σας αν θέλετε ή όχι. Η Επιτροπή πρόσθεσε το COP21 και τους κλιματικούς στόχους στην πρόταση ΕΦΣΙ 2. Κάποιες από τις τροπολογίες που προτείνονται δεν περιλαμβάνουν αυτές τις μνήες, αλλά τις μετακινούν στον ορισμό της προσθετικότητας. Διερωτώμαν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Ίσως θα έπρεπε να παραμένουν μεταξύ των γενικών στόχων των ε, έργων που θα πρέπει να στηρίξουν οι ευρωπαϊκές εγγύησεις. Επίσης, η ερώτηση για τις περιοχές και περιφέρειες της τροπολογίας 13-14. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό απαντήθηκε στις πρώτες σας απαντήσεις. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος της μικροδιαχείρισης από την πλευρά του Κοινοβουλίου, καθώς προσπαθούμε να πιέσουμε για να ε, πάρουμε και εμείς τη θέση που μας ε, οφείλεται στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Καλό είναι να είμαστε εδώ λίγο επιφυλακτικοί στις κοινοβουλευτικές μας πρακτικές. Για τον ορίζοντα 2020, για το ΕΦΣΥ και το διαδοχό του βλέπω να αντιμετωπίζονται νέες προκλήσεις λόγω του Brexit. Ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό και όσα δορυφορικά προγράμματα κινούνται γύρω από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό θα επηρεαστούν από το Brexit στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο πιεζόμαστε για το μέλλον. Τι επιπτώσεις θα έχει το ΕΦΣΥ 2 πώς μπορεί να επεκταθεί στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην ΚΟΕ τώρα. Από την ΕΚΟΝ εδώ ο κύριος Ντεμάζη, τον οποίο τον βλέπω. Α, ο κύριος Βιέγκας. Αντικαθέτω τον ε, Θάμπιο. Εντάξει. Ναι, δεν ε, υπήρχε κανείς από την μπάτζετ, οπότε εκπροσωπώ και τις δύο. Είμαι σκιώδης εισηγητής μαζί με τον ε, Φαμπιό Ντεμάζη για την έκθεση αυτή. Λοιπόν, να συνοψίσω τη δική μας θέση για το πρόγραμμα αυτό. Φοβερές επιφυλάξεις διότι η αρχή που διαπνέει όλο αυτό το πρόγραμμα είναι μια λογική που αναζητά να μιλήσει για χάσματα και λήψεις στην αγορά με στόχο να δοθούν περισσότερες βοήθειες και επιδοτήσεις στον ιδιωτικό τομέα Εμεί δεν καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει γράμμιση, Καταλαβαίνουμε ότι το δημόσιο θα παραμένει δημόσιο και θα θέλουμε δημόσιε επενδύσει με δημόσιο επενδυτικό πρόγραμμα. Όχι απλώ θα αφήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να παρέμβει. Εδώ συστηματικά αναζητούμε μέσα ώστε ο ιδιωτικό τομέα να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευση. Μιλάμε για αποτυχίες στην αγορά, για σημεία όπου υπάρχει ε, δυσκολίες στις επενδύσεις. Δεν συμφωνούν όλα αυτά με τα όσα ευαγγελίζεται η Επιτροπή, ούτε με τα όσα υποτίθεται διέπουν τη φιλοσοφία μας για την ε, ε, οικονομία της αγοράς. Και ότι αφήνουμε ελεύθερη την ιδιωτική πρωτοβουλία να αναζητήσει την κερδοφορία. Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια που στην ουσία θα επιδοτήσει τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους, ευνοώντας τις ε, εταιρικές σχέσεις δημοσιοποιητικού τομέα, με τη χρηματοδότηση έργων που θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα και χωρίς την ύπαρξη αυτού του προγράμματος. Αυτό που μας φαίνεται απαραίτητο να υπογραμμιστεί είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε καθόλου αυτήν την διάθεση να ξεφύγουμε μπροστά στον μακρινό μελλοντικό ορίζοντα. Όχι, γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη αυτέ οι επιβολίε που ανέφερα, που έρχονται από την πρακτική ζωή τη Πορτογαλία λόγου χάρη. Με αριθμού, με πάμπολα στατιστικά στοιχεία. Η Επιτροπή προβάλλει την Πορτογαλία ω την χώρα που έχει ωφεληθεί τα μάλλα από αυτό το πρόγραμμα. Εμεί στην Πορτογαλία τίποτα δεν έχουμε δει. Τι είχε γίνει από το ΕΦΣΥ. Ούτε μία επένδυση από το Δημαρχείο τη ε, Λισαβόνα. Ένα δάνειο των 50 εκατομμυρίων μόλι εγκρίθηκε από ε, το Δημοτικό Συμβούλιο τη Λισαβόνα υποτίθεται, αλλά αυτά είναι σενάρια. Σενάρια τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιβληθεί μια θετική εικόνα και να επιβληθεί και η παράταση αυτού του προγράμματος ε, καταπιεστικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση και ανάλυση όπως ε, ε, υπονοούσε και ζητούσε η πρώτη έκθεση που εγκρίθηκε από αυτό το κοινοβούλιο και την υποβολή του προγράμματος αυτού σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ήταν ένας από τους όρους. Έχουμε πνιγεί σε αυτή τη θάλασσα από αμφιβολίες και απορίες. Με την προσθετικότητα που αναφέρθηκε, τη γεωγραφική κατανομή, θέματα τα οποία από ό,τι φαίνεται από στατιστικής πλευράς έχουν ε, παραποιηθεί όσο περισσότερο γίνεται. Και ως προς αυτό η ιστορία επαναλαμβάνεται, διότι ήδη είχαμε ένα σύμφωνο ανάπτυξης και παρασταθερότητας το οποίο στην πρακτική είδαμε να μην μπορεί να καλύψει τις προσδοκίες. Οπότε που φτάσαμε τώρα σε αυτό το χρονικό σημείο, σημειώνουμε τις, θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις ε, αμφιβολίες και τις απορίες μας, αλλά βρισκόμαστε εδώ και περιμένουμε να μας πείσετε, μπας και αποδεχτείτε ότι δεν είχαμε δίκιο. Αλλά αυτές οι υποσχέσεις, αυτά τα σενάρια φαίνεται να λαμβάνουν σάρκα και οστά, παρά τις δικές μας αντιρρήσεις. είμαστε λοιπόν εδώ, αλλά χωρίς να σας χειροκροτήσουμε, ούτε να αναγνωρίσουμε τη βαθιά αξία αυτού του προγράμματος. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Έκχαουτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να παραμείνω στο δίλεπτο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους εισηγητές για τις προτάσεις τους. Βλέπω μια-δυο βελτιώσεις σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Νομίζω ιδίω όταν συζητάμε για το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπάρχει περιθώριο για ε, βελτίωση. Υπάρχει και το Διευθυντικό Συμβούλιο, το Steering Board. Εκεί επίση οι, τιμολο... οι αξίε τη τιμολόγηση πρέπει να αλλάξουν και να μην λαμβάνεται ως copy-paste το μοντέλο τη ΕΤΕ. Ε, επίση τα κριτήρια αιρεσιμότητας. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Αν σκεφτεί κανείς το ΕΦΣΥ, θα πρέπει να ξέρει ότι κάθε επένδυση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικού μας στόχους. Και δεύτερον, να γνωρίζουμε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, δεν θα ήταν εφικτό χωρί το εύση. Αυτό είναι η προστατικότητα. Εάν ε, κοιτάξουμε την τωρινή πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι λέει γι' αυτό, κάπως το βελτιώνει, αλλά στην ουσία δεν το βελτιώνει. Βλέπω και και ότι και οι συγκητέ πρόθεσαν να το επεξεργαστούν κάπω, αλλά δεν είμαι βεβαίω ότι με, όλε αυτέ τι πρόσθετε αλλαγέ δεν κάνουμε μια πρόταση τελικά όπου η προσθετικότητα και πάλι δεν καταλήγει να είναι ένα άδειο κέλυφο. Η αναφορά στους στόχου τη χιλιετία, λόγου χάρη που είναι τόσο ευρύ ο ορισμός τους που τι θα πούν. Εάν δεν προσέξουμε εν τέλει όλα θα εντάσσονται, θα είναι προσθετικά, ε, θα μπορούν να, να επιλεγούν. Στην ουσία δεν θα έχουμε κριτήρια επιλογή. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κριτήρια προσθετικότητα είναι πραγματικά προσθετικά ζωρευτικά. Να συνεισφέρει το ΕΦΣΙ στην επιτέψη των στόχων μα τα χρήματα που του δίνουμε και που θέλουμε να δαπανίσουμε, δεν θα πετύχει έναν τίποτα αν δεν υπήρχε το ΕΦΣΙ. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και να φανεί και από τι τροπολογίε μα. Ευχαριστούμε κυρία ότι Στα δύο λεπτά μείνατε στο παράδειγμα για όλου μα. Ελπίζω να το κάνανε όλο αυτό και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι και μα κάναν τη χάρη. Ο κύριος... προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχα τη δυνατότητα να πω ότι το ΕΦΣΥ είναι καλή ιδέα κατ' εμέ. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρακτική της εφαρμογή θα έπρεπε να βελτιωθούν κάποιες πτυχές. Έχουμε τώρα την πρόταση παράταση. Γι' αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να βελτιώσουμε ορισμένα σημεία. Το πρώτο, το είπε ο συνάδελφο ο Μπά, το θέμα τη προσθετικότητα. Η προσθετικότητα είναι προσθέμενη αξία ουσιαστικά αυτού του επενδυτικού προγράμματος και θα πρέπει να προστατεύσουμε ε, την αρχή αυτή. Να μην έχουμε το clouding out και επίσης ε, θα πρέπει να προωθήσουμε τα έργα εκείνα τα οποία στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν αστοχίες στην αγορά, γιατί έχουμε πρόβλημα όχι τόσο ρευστότητα ε, στην έλλειψη επενδύσεων, ε, όσο επένδυση ε, σε ρηψοκίνδυνα έργα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί μπορεί να παίξει ρόλο λοιπόν αυτό ο παράγοντα τη σε Ένα δεύτερο σημείο. Περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη πληροφόρηση, ενημέρωση, υποχρέωση για πληροφόρηση, ιδίω ε, σε ό,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και όλα αυτά βέβαια σημαίνουν ότι θα πρέπει και οι εκθέσεις αξιολόγησης ε, από την Επενδυτική Επιτροπή να είναι προσβάσιμες για να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τρίτο σημείο, τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από εδώ και πέρα με το ΕΦΣΙ 2.0 μπορούν να πάνε εκεί που δεν είχαμε φτάσει μέχρι τώρα. Κοινωνική υποδομή, περιβαλλοντικά έργα, ενεργειακή απόδοση, μικρότερης κλίμακας έργα. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε να διευκολύνουμε τη δημιουργία επενδυτικών πλατφορμών, γιατί για μικρή κλίμακα έργα αυτή είναι η μόνη δυνατότητα πρόσβαση στη χρηματοδότηση του ΕΕ. σε Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για το EFTT έχω τον Μαρκοβάλη στο καταλογό μου, αλλά δεν τον βλέπω. Υπάρχει κανείς από το EFTD, ουδής από το ENF, Μάρκο Τζάνι. Τι έγινε. Και αυτός έφυγε. Πήραν τη και δεν είναι το ένας αυτό το άλλος. Μα υπάρχει κανείς από τον επίσημο κατάλογο, όχι. Άρα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδες εισηγητές που τήρησαν το χρόνο αγόρευσης και ξαναδίνω τη σκητάλη στον πρόεδρο της Επιτροπής Προεπιλογισμών για τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Ευχαριστώ. ΚΑΤΣΔΙ λοιπόν. Κύριε Μπερές. Ευχαριστώ. Καλύτερα από την προηγούμενη φορά, γιατί δεν είχαμε καρδιά την προηγούμενη φορά. Είναι σημαντικό να έχει ο καθένα την ευκαιρία να μιλήσει. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τον εισηγητή. Δύο-τρία ζητήματα από του εισηγητέ που προέβαλαν τα δύο-τρία θέματα στο λίγο χρόνο που είχα στη θέσή του. Πώ το έτσι καταρχά συνδυάζεται με τους, ε, διαμεσολαβη... τους ενδιάμεσους τους ε, παράγοντες εκείνους που μπορεί να είναι οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην κάθε ζώνη ενδιαφέροντος ή στο κάθε τόπο ε, και άλλα θέματα στα οποία θέλω να αναφερθώ αλλά δεν έχω τόσο χρόνο θα τονίσω λοιπόν τρία ζητήματα καταρχάς αυτό που βλέπουμε στα κράτη-μέλη και διάρθρωση με τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν συμμετάσχει, δεν έχουν συμβάλει στο έτσε. Την ώρα που εμείς αγωνιζόμασταν για να εξασφαλίσουμε την δική τους την επένδυση και με το όφελος της ευελιξίας που μας εξασφάλιζε η ανακοίνωση της Επιτροπής. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το αλλάξουμε, να βελτιώσουμε δηλαδή το βεληνικές του έτσε. Δεύτερο, τροπολογία υπαριθμών 2 και νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία επικαλούνται οι εισηγητέ στο πλαίσιο τη αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ήθελα πιο πολλέ λεπτομέρειε και διευκρινήσει εκ μέρου των εισηγητών, αλλά θα επανέλθω στο κύριο ζήτημα, ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Ο κύριο Στόρβαλτ, ο κύριο Ινκούτ επίση τοποθετήθηκαν προ την ίδια κατεύθυνση. Σημειώνω. Δηλαδή, Ε, προσπαθώντας να υλοποιήσουμε το στόχο των ΗΠΑ την Ατζέντα για την Ανάπτυξη και εγκαταλείποντας τη στόχευση σαν όρο του 40% για τους στόχους της COP21, ε, ε, μήπως κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα, μήπως κινδυνεύουμε να χάσουμε τον μπούσουλα. Καταλαβαίνω ότι η βασική ιδέα είναι πως προσπαθούμε με περι... να... να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση, με καλύτερη χρηματοδότηση για, τα κοινωνικά, για τις κοινωνικές επενδύσεις κτλ. Αλλά πρέπει να δούμε κιόλα επιτυγχάνονται οι στόχοι. Τη COP21. Εγώ για το έτσι... Είχα αγωνιστεί, όπως και με τους συναδέλφους Επιτροπής Βιομηχανίας, Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχαμε αγωνιστεί λοιπόν να εξασφαλιστεί η ρητή στόχευση στους στόχους αυτούς και συγκεκριμένοι πόρη αφιερωμένοι στους στόχους αυτούς. Με ανησυχεί λοιπόν το γεγονό ότι ανοίγει πάλι αυτή η συζήτηση. Και ναι, καλό είναι να έχουμε μια ευρεία στόχευση, αλλά παρόλα αυτά δεν θα ήθελα να χαθούν αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Τζιλ. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να καλωσορίσω την έμφαση που διατυπώνει ο εισηγητής σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε ελλείμματα, ε, ελλείψεις σε πολλά σημεία και ιδιαίτερα αυτά που ε, ανέφερε και η Περβάνος Περές αναφορά στην κλιματική αλλαγή, COP21. Βέβαια δεν θα σε ακολουθήσω μέχρι τέρμα σε αυτά που είπες Περβάνος, αλλά είναι σημαντικό να είναι σαφής αυτή η εικόνα, αυτή η διάσταση. Κύρια επίκριση από πλευρά μου είναι αυτή που καλύπτει η τροπολογία 29 του εισηγητού που διορθώνει, αποκαθιστά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει φαίνεται την ε, δεδομένη την εικόνα ότι είναι άντρες όσοι διατυπώνουν προτάσεις. Μια πρόταση λοιπόν της Επιτροπής δεν μπορεί να έχει αυτή τη διατύπωση. Για το έτσι, χρειαζόμαστε καλύτερη δομή διακυβέρνησης, διαχείρισης. Επίσης χρειάζεται το έτσι να υποστηρίζει όλες τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές σε όλη την Ένωση και να, έχει περισσότερη, να δίνει περισσότερη έμφαση στη στέγη και άλλους τομείς, κοινωνικές δομές και όχι μόνο παραδοσιακές μορφές επενδύσεων. Ξέρω ότι προσπάθησε ο εισηγητής να τα καλύψει όλα αυτά, αλλά όσο και αν τα θεωρώ ευπρόσδεκτα όλα αυτά, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, στην διατύπωση των προτάσεών τους, να μην ε, αναφέρονται μόνο σε αρσενικό γένος. Ο κ. Μαυρίδης. Ε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η όποια κριτική δεν σημαίνει αντίθεση με το ίδιο το ΕΦΣΥ. Και ε, γι' αυτό και έχουμε προτείνει, έχουμε υποβάλει αρκετές προτάσεις που θεωρούμε ότι βελτιώνουν το όλο project. Ε, για παράδειγμα, διασυνοριακή συνεργασία με τρίτα κράτη-μέλη. κράτη, είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουμε. Δεύτερο, φρέσκο χρήμα και όχι από τα υφιστάμενα προγράμματα. Δεν συνενούμε στην αντικατάσταση των Ταμείων Περιφερειακής Πολιτικής. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να επικεντρωθώ είναι το εξής. Κατ' εμέ υπήρχε μια προσδοκία ότι από το ΕΦΣΥ θα υποφελούνταν συγκριτικά, other things being equal, περιοχές και κράτη που πλήγηκαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Κοιτάζοντας τη γεωγραφική κατανομή, νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνει πως το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχαμε αρχικώς. Και θα κλείσω με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Συμμερίζομαι την άποψη ότι το country profile και το risk profile είναι δύο στοιχεία που μπορεί να διαφοροποιούνται τόσο πολύ που να κάνουν ένα έργο αποδεκτό ή ένα έργο μη αποδεκτό. Είναι γι' αυτό που επιμένουμε ότι για μικρά κράτη-μέλη, όπως και η Κύπρος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους, ένα τέτοιος είναι το blending του ΕΦΣΙ με επιδοτήσεις, ούτω ώστε μικρά κρατημέλη με πολύ ψηλό country risk να μην υποφέρουν από αυτό που ονομάζω εγώ ως exclusion bias, επειδή τελικά απορρίπτονται έργα που σε άλλα κράτη θα γίνονταν αποδεκτά. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό και είμαι βέβαιος ότι το συμμερίζονται και πάρα πολλοί άλλοι. Σας ευχαριστώ. La parole est maintenant à Monsieur Roux. Κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να τονίσουμε ότι το σχέδιο Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων, το Juncker Plan όπως επωνομάζεται, είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων από καταβολή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να το μηδενίζουμε. Ποτέ άλλοτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρξε μια ανάλογη επενδυτική πρωτοβουλία. Και από αριστερά μέχρι δεξιά όλοι διαμαρτύρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν κάνει επενδύσει και δεν αναλαμβάνει επενδυτικέ πρωτοβουλίε. Ιδούν μια τεράστια επενδυτική πρωτοβουλία. Και θα πω ότι η σημαντική συμβολή για να έχουμε αυτή τη σημαντική επενδυτική πρωτοβουλία την έχει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ δεν πρέπει να μηδενίζουμε την προσπάθεια, ιδιαίτερα των δύο αγαπητών εισηγητών, του κ. Φερνάντε και του κ. Φούλμα, που χωρί τη δική του μεγάλη σημαντική θετική συμβολή, το ΕΦΣΙ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα έστω με τα προβλήματα και τι δυσκολίε. Βελτιώθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν όταν ήταν αρχικά ο σχεδιασμό αυτού του ΕΦΣΥ και το ότι σήμερα συζητούμε για τροποποίησει είναι σημαντικό γιατί υπήρξε πρωτοβουλία από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Μια τέτοια τεράστια επενδυτική πρωτοβουλία θα ήταν πραγματικά ε, θα ήταν μαγικό να μην υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το σημαντικό πρόβλημα έγκυται στο ότι μικρέ και αδύνατε οικονομικά χώρε φαίνεται ότι δεν έχουν την ευχαίρεια να πάρουν αυτά τα προγράμματα και να επενδύσουν. Είτε γιατί είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο που βγαίνει μέσα από, τον, από την θέση κινδύνου αυτή τη χώρα, είτε για άλλου λόγου. Και οφείλω να πω ότι από τη δική μου εμπειρία, η Κύπρος που δοκιμάστηκε και πέρασε μέσα από μια οικονομική κρίση, που έπρεπε να είναι από τι χώρε που θα μπορούσαν να πάρουν μερίδιο από αυτήν την μεγάλη σημαντική επενδυτική πρωτοβουλία για να μειώσει και την ανεργία τη, για να δώσει νέε θέσει εργασία, για να δημιουργήσει νέα ανάπτυξη, για να δημιουργήσει όθηση, δεν μπόρεσε να πάρει ουσιαστικά ούτε ένα έργο. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το ζήτημα και να βρούμε λύση. Δεν είναι μόνο γεωγραφική κατανομή. Πιστεύω ότι το ΕΦΣΙ θα μπορούσε να ήταν ΕΦΣΙ δύο ταχυτήτων. Δηλαδή των πολύ προηγμένων ανεπτυγμένων χωρών που ήδη αναπτύσσουν από μόνοι τους επενδυτικέ πρωτοβουλίες τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή από μόνε τους οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδύσει, και οι άλλες χώρες που είναι αδύναμες και δεν έχουν αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τι επενδύσει, πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορετικά κριτήρια κίνητρα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν αυτή τη μεγάλη επενδυτική πρωτοβουλία που τιμά την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει έργο και η Ευρώπη για επενδύσει και για του πολίτε. Ευχαριστώ. Merci. Madame Ευχαριστούμε κυρία Μάλετιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι στην αρχή όταν εισήγαμε το ΕΦΣΥ μιλούσαμε για τρεις πυλώνες και ένας από τους πυλώνες ήταν τα προγράμματα Ready to Go και Project Pipeline. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε με προσοχή όλα τα επενδυτικά προγράμματα. Υπ' αυτήν την πρόκτικη. τα ready to go, τα έτοιμα δηλαδή να εκτελεστούν και τα, ε, τους διάβλους προγραμμάτων και έργων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δει πώς αντιμετωπίσει το πρόβλημα κάποιων χωρών όπου οι τράπεζες λένε ότι οι μικρομεσαίες δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια. Θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες. Αυτό θέλουμε να γίνει και να πείσουμε τους ε, μεσάζοντες, τράπεζες και άλλους ενδιαμέσους πώς μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ της ΕΤΕ και των μικρομεσαίων. Σας ευχαριστούμε. Φτάνουμε στον κατάλογο αυτής της διαδικασίας του Catch the Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα αιτήματα Τώρα, ερωτήσεις προ τους εισηγητές. Οι μικρομεσαίες θα πρέπει να έχουν και λιγάκι διάθεση κατακτητική, να επεκταθούν και σε ε, αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εδώ, οι εισηγητέ βλέπουν τη δυνατότητα να δοθούν δάνεια σε μικρομεσαίε που θα παρουσίαζαν ένα σχέδιο έργου ή προγράμματο με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, με αυστηρή πλαισίωση για να προσπαθήσουν να κατακτήσουν αγορέ εκτό πλαισίου Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριοι εισηγητέ, θα έχετε τώρα τη δυνατότητα να εκφραστείτε. Ποιο θέλει το λόγο πρώτο, Ο κύριο Μπούλμαν ή ο κύριο Φερνάντε, Ο κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πλήρη συνεργασία και απόλυτα διαφανώς βλέπετε ότι λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ερώτημα, ναι, αν είναι προσθήκη. Η χώρα μου έχει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την ε, διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα είμαστε μπροστά και νομίζω ότι εκεί ε, μπορεί να δραστηριοποιηθούν περισσότερο τα διαδοτικά ταμεία. Για το ΕΦΣ πιο πολύ θα έλεγα ότι έχει στόχο τις επιχειρήσεις. Να προσπαθήσω τώρα να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα. Τροπολογία 2. Γιατί. Διότι θέλουμε να συνεχιστεί το ΕΦΣΙ και γιατί είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένο με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το ΕΦΣΙ. Ουσιαστικά η εγγύηση της χρηματοδότησης είναι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και δεν είναι τυχαίο ότι το δεύτερο ΕΦΣΥ ε, πηγαίνει μέχρι το 2020. Δεν ξέρουμε αν το επόμενο πολιτές σωμικό θα φτάσει μέχρι το 2025, 2024, 2026 κτλ. Αλλά θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το 2020 να μπορεί να καταθέσει μια νομοθετική πρόταση ώστε να συνεχιστεί το ΕΦΣΥ. Υπάρχει κάτι σημαντικό εδώ. Υπάρχουν πολλά έργα για τα οποία απαιτείται μακροχρόνια προετοιμασία. Χρειάζεται λοιπόν προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια λοιπόν στο ΕΦΣΙ γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για πιο μεγάλης κλίμακας έργα, παράδειγμα χάρη, για τις ε, πλατφόρμες μεταξύ χώρων, τις διασυνοριακές πλατφόρμες. Είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιες πλατφόρμες διασυνοριακές πλατφόρμες. Υπενθυμίζω, η Ένωση της Ενέργειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, αλλά με πλατφόρμες που έχουν αυτό το στόχο. Με τρίτες χώρες θα ήταν πολύ σημαντικό για να μην εξαρτώμεθα όπως εξαρτώμεθα σήμερα. Επί παραδείγματι από τη Ρωσία. Αυτά ως εξήγηση για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Το λόγο ταμείο μας υποχρεώνει να είμαστε προβλεπτικοί, proactive όπως λέμε στα αγγλικά και να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Ουσιαστικά δεν παίρνει χρήματα από τα διευθυντικά ταμεία. Μπορεί να βοηθήσει την εκτέλεση και ουσιαστικά να προσφέρει μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ γραφωτικών ταμείων και αυτού του ταμείου. που πολλές φορές το λέμε σχέδιο Juncker. Και υπάρχουν επενδύσεις, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, που δεν μπορούν να τις πραγματοποιήσουν, ε, τα διευθυντικά ταμεία μπορούν μόνο κατά μέρο να ε, πραγματοποιήσουν την ελόγω επένδυση, αυτό το ταμείο έρχεται συμπληρωματικά, προσθετικά. Και πρέπει και μπορεί να το κάνει. Συμφωνούμε πάνω σε ένα πράγμα. Μεγαλύτερη διαφάνεια και ορατότητα για αυτό το ταμείο, έχει βοηθήσει ήδη πολλές ΜΜΕ, αλλά πολλές φορές δεν το γνωρίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρουν καν ότι έχουμε την εγγύηση του υπερπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις επενδύσεις. Εξίσου σαφές είναι ότι το Advisory Hub, αυτός ο συμβουλευτικό κόμβος, αυτό το κέντρο, πρέπει να βελτιωθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε και τις περιοχές εκείνες που δυσκολεύονται περισσότερο σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των έργων. Αλλά και σε προημότερο στάδιο, εκτέλεση ή δημιουργία πλατφορμών ή υποβολή υποψηφιωτήτων, κατάρτιση υποψηφιωτήτων. Περιμένουμε λοιπόν τις τροπολογίες σας. Υπάρχει και κάτι άλλο, με βέβαιος ότι θα τα βρούμε με τη συνάδελφο που δεν είναι τώρα εδώ. Για μας είναι σαφές ότι το ΕΦΣΙ θα πρέπει να σέβεται όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τις συμφωνίες και τη Συμφωνία των Παρισίων πόσο μάλλον. Και τα έργα που θα χρηματοδοτούνται θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Πού άλλου θέλω να επιμείνω. Σημαντική προσθετικότητα, αλλά δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν είναι το ρίσκο και ο κίνδυνο ο ίδιο παντού. Ούτε σε όλα τα κράτη-μέλα και μέσα στο ίδιο κράτο μέλο δεν είναι ίδιο ο κίνδυνο, το ρίσκο σε όλε τι περιοχές. Κοινωνικές επενδύσεις, είπατε είναι σημαντικό για τι κοινωνικέ υποδομέ. αλλά πρέπει να έχουν ρίσκο. Άρα, διαρωτώ με εγώ, μπορούμε να επενδύσουμε τελικά σε κοινωνικέ υποδομέ υπό αυτήν την έννοια. Το ΕΦΣΙ ήδη τώρα επιτρέπει την πραγματοποίηση επενδύσεων στο κοινωνικό τομέα. Και όταν μιλάμε για τα διαθροτικά ταμεία, προσοχή, οι συμφωνίε εταιρική σχέση δεν είναι ίδιες. Να δούμε την συμφωνία εταιρική σχέση με την Πορτογαλία, για παράδειγμα δεν μπορούμε να φτιάξουμε καμία σχεδόν υποδομή. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε αυτοκινητοδρόμους ή οδικό δίκτυο με τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στις χώρες εκείνες όπου τα διαρθρωτικά ταμεία δεν διευκολύνουν ή δεν μπορούν να καλύψουν επενδύσεις σε υποδομές, να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο. Η δεν μπορουν να καλυψουν επενδυσεις σε υποδομε να εχουμε λοιπον τη δυνατοτητα σε αυτε τι χωρε να αξιοποιησουμε αυτο το εργαλειο η πολιτικη συνοχης πρέπει να την δούμε με διαφορετικό μάτι και όχι με βάση το ρίσκο. Τώρα, είναι σφάλμα να ζητήσουμε ποσοστώσεις για το ΕΦΣΥ και ιδίως για τις χώρες συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε την ταφόπλακα στην πολιτική συνοχής. Και δεν είναι αυτός ο στόχος μας βέβαια, σε καμία περίπτωση. η Κομισιόν πρέπει να βοηθήσει και αυτή. ώστε αυτό το ταμείο να αξιοποιηθεί από κοινού με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και σίγουρα είναι απαραίτητες οι συνέργειες. Επίσης, ένα άλλο σημείο. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των πολιτικών ε, συνοχής. Αν μια χώρα ε, παίρνει επιδοτήσεις, ε, Πρώτα βλέπει τις επιδοτήσεις και μετά θα δει τα δάνεια. Ίσως και αυτό είναι μια εξήγηση που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και εγώ και ο Σαλφος Μπούλμαν που θέλω να τον ευχαριστήσω. Ε, περιμένουμε τη δική σας βοήθεια. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Το steering board λέμε ότι θα πρέπει να έχει εκπρόσωπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην είναι βουλευτής. Το θέμα είναι οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου να ενσωματωθούν στις κατευθυντήριες γραμμές. Θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριος Μπούλμαν. to... Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που αφού σε αυτήν την ε, συζήτηση. για την προσφορά αυτών των τόσο λεπτομερών πρέπει να ομολογήσω γνώσεων επίσης. Είναι άλλωστε η δεύτερη φορά που ασχολείστε πολύ από εσά με τα θέματα αυτά και βλέπουμε τους καρπούς της εμπειρίας σας, αλλά και για τους πιο καινούριου στην ομάδα. Ευχαριστώ ιδιαίτερως για την προσήλωση στον αγορά να εξασφαλίσουμε κάτι θετικό. Εξαιρετικά θετικό για μένα ως συνεισηγητή είναι προς, την, προς το παρόν ότι όσο, περι, όσο λιγότερο συμφωνούμε για το τι πρέπει να γίνει με το έτσι δύο ή τι θέλουμε να επιτύχουμε επί της ουσίας, τόσο την ε, συζήτησή μας την καθοδηγούν ε, τα μελήματα για την εξασφάλιση της κατάλληλης τεχνολογίας για την επιτεύξη των στόχων αυτών και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει και αποτελεί και επιβεβαίωση της ενότητας που έχουμε άλλωστε και στο παρελθόν επιδείξει. Ότμαρ. Ότμαρ και όχι η πρώτη φορά, επισημαίνει πολύ σωστά τι σημαίνει ορόσημα. Μας λέει θέλουμε να είμαστε στο Champions League. Βεβαίως. Το προσυπογράφω. Θέλουμε δηλαδή ένα καλής υψηλής ποιότητας έργο με το οποίο θα μπορούμε να πούμε «Να, δες τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση» και πάνω σε αυτό να μπορούμε να στηριχθούμε και να προβάλλουμε όχι μόνο την ποσότητα αλλά και την ποιότητα. Ρητά αποστηρίζω αυτή την προσέγγιση, συμφωνώ απολύτως. Και εδώ εγγράφεται και το πάγιο επιχείρημά του, ότι δεν πρέπει να χανόμαστε ούτε σε περατιολογικές δομές, ούτε σε αυτό που θα ονόμαζα εγώ πυλωνοποίηση, δηλαδή ποσοστός επί ποσοστός, επί ποσοστό. Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό δεν είναι το ίδιο με το να προσπαθούμε το έτσι ή κάποια σημαντικά του τμήματα να το μετακινούμε προς τους ε, βιώσιμους στόχους για την υλοποίηση κάποιων έργων. Ξέρω ότι άλλοι και ιδιαίτερο Εμμανουέλ θα ασχοληθούν με την ε, δημοσιονομική διάσταση κυρίως στον προπολογισμό. Προσβλέπω στην υποστήριξή τους, όπω και των λοιπόν συναδελφών τη Επιτροπή των Προπολογισμών, που ξέρουν πολύ περισσότερο από ό,τι οι συναδελφοί τη ΕΚΟΝ, τι είδου συνέπειε μπορεί να έχει το ΕΤΣΕ στον, για τον προπολογισμό και ιδιαίτερω είναι εξοικειωμένοι με την ε, πληθώρα και ποικιλία ιδιαίτερων συνθήκων που μπορούν να επικρατούν σε διάφορε περιοχέ και περιφέρειε. Και επίση, μιλούμε για ευφυή συνδυασμό κονδυλίων των διαρροτικών ταμείων με του ΕΤΣΕ χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα απορροφηθεί από τη νέα τεχνολογία έτσι το ε, διαρθρωτικό ταμείο. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο, να παραμένει ανεξάρτητο ως μέσον και για την εξυπηρέτηση των έργων του έτσι, στη τελευταία ανάλυση. Σάντερ, ιδιαίτερα σημαντικά τα σχόλιά σου και την προηγούμενη φορά και τώρα. Τα βρίσκω πολύ επικοδομητικά. Οι συνεισηγητές ήδη προσπάθησαν να ε, λάβουν υπόψη τα πορίσματα Ernst Young και αναζήτησαν λύσεις για crowding out, για αναζήτηση ιδιωτικών πόρων, που όμως δεν μπορεί να είναι η πρόθεση του έτσι. Θα θέλαμε να δούμε συγκεκριμένες προσεγγίσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές δυνατότητες σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, με προσοχή παρακολουθήσαμε τα όσα υποδεικνύει το ελεγκτικό συνέδριο, σωστά επισήμανες, ότι είχε αρχικά προβλέψει ένα πιο χαλαρό χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται άλλωστε για έναν από τους λόγους για τους οποίους αφενός ως συνεισηγητές, ο Χωσέ Μανουέλ και υποφαινόμενος, είπαμε ότι έχουμε σαφή στόχο, εκπεφρασμένη βούληση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Μάλτας να το ολοκληρώσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αφήσουμε επαρκή χρόνο για μια υγεία συζήτηση στην υπόθεση αυτή, γιατί τον χρόνο τον έχουμε. Ούτε μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν ε, είναι εν εξελίξη το έτσι, δεν λειτουργεί εντωμεταξύ, ότι δεν έχει πόρους να διαθέσει. Νίλ Στόρμαρς. Ο Νίλς μας επισήμανε τον κίνδυνο να παραγνωριστούν τα επιτεύγματα της Επιτροπής σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Δεν ήταν στόχος μας αυτό. Αυτό το είπε και ο Μπάρς Πράσινη συναδελφή από τους προπολογισμού. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την διαφύλαξη της προσθετικότητας, της έννοιας, της διάστασης, της ποιότητας. Αυτή ήταν και η πρώτη θέση μας εξ αρχής, δηλαδή να, να διαφυλαχθεί αυτό, αλλά και να συμπεριλάβουμε και την κοινωνική διάσταση, που ήδη προβλεπόταν ε, και για το έτσι ένα, αλλά δεν έχουν ληφθεί υπόψη σημαντικά έργα από τον κοινωνικό ε, τομέα στο έτσι ένα, Το λαμβάνουμε λοιπόν και αυτό. Σάντερ, Μπέντ, ECR ε, επισήμαναν την ε, αναγκαιότητα της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, την βελτίωση του ίδιου χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τις τεχνικές και καλούμε και τους πράσινους συναδέλφους ε, επίσης να συμβάλλουν στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο διαχείρισης, αν είναι καλές οι προτάσεις, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να τις λάβουμε υπόψη και να τις ενσωματώσουμε και σε ε, συμβαστικές τροπολογίες. Είναι να έχει αποχωρήσει, πάντως σημειώνω ότι συν οι συγητές έχουν εξουδετερώσει την αναφορά πάντα σε αρσενικό γένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας μην ανησυχεί η κυρία Τζιλ. Για τον κύριο Μαυρίδη. Αναφερθήκατε στα περιφερειακά ταμεία. Είπατε ότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το διαφορετικό προφίλ κινδύνου του κράτους μέλους. Ο κύριος Χριστοφόρου υπεγράμισε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα, η ιδιαίτερη κατάσταση στην Κύπρο. Και στις περιφερειακές δομές ο κύριος Μαυρίδης μας είπε, που ανέφερε ο κύριος Μαυρίδης, είναι, αφορά και τις δύο πλευρές. Ο Χωσέ Μανουέλ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχουν καλά hub, αποτελεσματικά hub και να ενισχυθεί το δυναμικό η ανάπτυξη δυναμικού, το capacity building. Χωρίς αυτό και τα hubs δεν μπορούμε να έχουμε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε, έχει επισημάνει και η κυρία Μάλετιτς. Βεβαίως θα προσπαθήσουμε όλα τα θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, με την υποστήριξη σας ελπίζω, να τα αναπτύξουμε και θα σας πούμε πού ακριβώς χρειαζόμαστε βοήθεια από πλευρά σας για τη διατύπωση των τροπολογιών. Πρόεδρε, ναι, οι μικρομεσαίες έχουν δικαίωμα να επενδύουν, πρέπει να έχουν ε, την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σωστό το βρίσκω αυτό, αλλά μπορούν ε, να εξάγουν έργα να βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο Ότσμαρ, θα ήθελα και εγώ περισσότερα διασυνοριακά έργα και εγχειρήματα, ώστε να τονιστεί και το διεθνές μας προφίλ, αλλά και η διασυνοριακή, η ευρωπαϊκή διάσταση της, των επενδύσεων μας. Ευχαριστώ πολύ και ε, παρακαλώ να λάβετε υπόψη ότι οτιδήποτε έχετε να προτείνετε είναι ευπρόσδεκτο. Ε, περιμένουμε τις ιδέες σας, θα τις ε, δεχθούμε ε, με θετικό πνεύμα. Θέλουμε συνεργασία, άλλωστε αυτή είναι και η δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συνεργασία όπως και στο προηγούμενη φορά άλλωστε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον εισηγητή και τον Σκιώδη. Και όσους πήραν το λόγο για να τοποθετηθούν, η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Απλώς μια παρατήρηση προσωπική για τα προγράμματα έργα με κοινωνική διάσταση. Είναι ένας από τους στόχους, αλλά στην ουσία τι είναι ένα πρόγραμμα με διάσταση κοινωνική που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΥ. Δεν είναι και τόσο απλό να το ορίσουμε. Πώς μπορεί ένα έργο να θεωρεί ότι θα προσφέρει κέρδος αποπληρώνοντας το δάνειο που δόθηκε. Δημιουργώντας τέσσερις απασχόλησης και δυναμικά, οικονομικά μάλλον δυναμικό χαρακτήρα. Δεν είναι και τόσο προφανές. Να σας ενημερώσω τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 9ης Ιανουαρίου και 13ης Φεβρουαρίου σας έχουν αποσταλεί. Έχετε λάβει γνώση και δεν έχουν υπάρξει παρατηρήσει από την πλευρά σας. Ε, άρα θα εγκριθούν. Δεν ακούω να υπάρχει, κανείς, να υπάρχει αντίρρηση από κάποιον. Εν τω μεταξύ, η Προεδρία της Μάλτας ελπίζει να ολοκληρωθεί αυτή η νομοθετική πορεία στην ευεία εξαμήνου τη και έχουμε πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Οι τροπολογίες για τα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο. Την Τετάρτη 23 Μαρτίου, με συγχωρείτε, την Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα, 23 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα, θα συζητήσουμε στις 3 Απριλίου ταυτόχρονα το σχέδιο έκθεσης και την έκθεση εκτέλεσης και θα ψηφίσουμε σε κοινή συνεδρίαση της των Επιτροπών ε, Μπούτς και ΕΚΟΝ στις 24 Απριλίου. Για το σχέδιο έκθεσης και για την έκθεση εκτέλεσης. Υπάρχουν άλλε ερωτήσει ή παρατηρήσει. Όχι. Σα ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τη συμμετοχή σα. Ε, κυρίω τη λήξη τη συνεδρία.